για τις σχέσεις με τις χώρες Μαγκρέμπ. Υπάρχουν σχόλια, παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος το λόγο. Θεωρώ λοιπόν ότι έτσι εγκρίνεται αυτός ο διορισμός.